Bonjour Καλή σας μέρα. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Γι' αυτό παρακαλώ ας κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν οι κάρτες μας ε, λειτουργούν καλά. Δοκιμή λοιπόν. Ξεκινάει η ψηφοφορία, αυτή η δοκιμαστική δηλαδή. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Βάλτε τις κάρτες σας παρακαλώ για να δούμε αν ε, λειτουργούν καλά. Είναι 7 που δεν έχουν ψηφίσει. Άλλοι δύο παρακαλώ να ψηφίσουνε. Πέραστη της ψηφοφορίας. Ε, εντάξει είναι. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία του Μηχανισμού Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Εγκρίνουμε την έκθεση του κυρίου Μίτσελ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, οπότε ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Δεν δούλεψε το μηχάνημα. Για δοκιμάστε σε κάποιο άλλο. Καθίστε κάπου αλλού καλύτερα. Ο κύριος Κλίντσι μπορεί να αντικαταστήσει τον κύριο Βάγκελε γιατί είναι ένας παραπάνω έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν υπάρχει θέμα, μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά. Εντάξει, ψηφίσατε όλοι. Τώρα κλείνει η ψηφοφορία. Και ψηφίστηκε υπέρ ομόφωνα. 29 ψήφοι υπέρ. Συνεχίζουμε. Και περνάμε στα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Έκθεση Γκέρενς. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες Ψήφισαν 28 υπέρ και μία αποχή. Τώρα ψηφίζουμε για την φορολογία και ανάπτυξη. Τροπολογία 27. Μπορούμε να ψηφίζουμε, παρακαλώ, λέει ο κύριος Μπέρμαν, unblock όσο γίνεται περισσότερο, γιατί η έκθεση αυτή έχει πάρα πολλές τροπολογίες. Όπου μπορούμε λοιπόν, unblock, παρακαλώ. Όχι, φοβάμαι ότι θα είναι περίπλοκο αυτό, λέει η Προεδρο. Λοιπόν, τροπολογία αριθμό 27. Ηλεκτρονικά, εντάξει, είναι πιο απλό. Λοιπόν, ηλεκτρονικά τα πάντα. Παρακαλώ, κύριε Μαρτίνεθ. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Μαρτίνεθ, δεν τον ακούμε. Δεν ακούγεται ο κύριος Μαρτίνεθ, δεν έχει πατήσει το μικρόφωνο του. Διαμαρτύρεται, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Μα δεν είναι δυνατόν 100 τροπολογίε να τι ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό, λέει ο κύριο Μαρτίνεθ. Πρόεδρο. Εντάξει. Διανατάσσεω τη χειρό. Και όταν θέλει κάποιο επαλήθευση, τότε θα επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Η τελική ψηφοφορία όμω θα γίνει ηλεκτρονικά. Σύμφωνοι. Ωραία. Ωραία. Τροπολογία 27. Υπέρ παρακαλώ. Διανατάσσεω χειρό. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα, Ρυθμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 καταπίπτει. Οπότε πάμε τώρα στην τροπολογία της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Υπέρ παρακαλώ. Η 4 ήταν. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία ΙΝΤΑ. ρυθμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ίντα 9. Είναι κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα παρακαλώ. Χωρίς το θετικό υπέρ. Κατά. Αποχές. Εδώ θα επαληθεύσουμε. Οπότε ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Μία ψήφο λείπει. Α, εντάξει τώρα. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου του κύριου Μίτσελ. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα, συμβαστική τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 34, 35 και 36 καταπίπτουν. Και έτσι Περνάμε στην τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία σε τώρα, γάμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42, όχι. Φτάνουμε στη 45 έτσι, με κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία ίντα. Δύο κατατμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα, ντε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 1 τώρα. Με κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο κύριος Μίτσελ. Κύριε Πρόεδρο, για την διατύπωση της συμβαστικής, εγώ κατά κατάλαβα ότι είχε αλλάξει η ορολογία όσον αφορά το τάξ. Είχαμε συμφωνήσει. Η γραμματεία λέει ότι έχετε δίκιο και ότι όντως έτσι είναι. Συμβαστική τροπολογία ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53, καταπίπτει. Φτάνουμε στην 56, έτσι. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, κύριε Μίτσελ, για την 58, μισό λεπτό να βάλω τα ακουστικά μου, λέει ο πρόεδρο. Για την 58, κύριε πρόεδρε. Για να είμαστε συνεκτικοί ανάμεσα στην 158 και την 58. Στο δεύτερο τμήμα, στο σίγμα F, που μιλάει για την ε, επαλήθευση στον αφορά τον εταιρικό φόρο κτλ. να είναι ακριβώς η ίδια διατύπωση όπως και στο 58 και χωριστή κατά τμήματα ψηφοφορία να γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ψηφίζουμε πρώτα σε κατά τμήματα ψηφοφορία την ε, προφορική 2 υπέρ, το πρώτο, κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ Μια στιγμή. Ένας-ένας. Ο κύριος Κλίντς καταρχήν που είναι ο συντάκτης της τροπολογίας αυτής. Θα ήθελα να τροποποιήσω την προφορική τροπολογία για γλωσσικούς λόγους, παρακαλώ. Και θα ήθελα αντί να λέει by the calculation, να λέει by calculating κτλ. Αντί να λέει by the calculation of income tax rates. Μάλιστα, με την τροποποίηση αυτή δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε 58 καταπίπτει και περνάμε στην ίντα 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ίντα 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 60. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κύριε Μίτσελ, κύριε Πρόεδρε, το ΕΛΚ δεν συμφωνεί με την προφορική τροπολογία αριθμός 3 και θα και για την 4 για να κερδίζουμε χρόνο. Καλώς. Οπότε δεν ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία 3 και ψηφίζουμε την 63 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η προφορική 4 είπαμε ότι καταπίπτει, γιατί δεν συμφωνείτε. 65. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Ψηφίστε λοιπόν γιατί είναι 65 ηλεκτρονικά. Ξεκινήστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία σιγματάφ. F υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 71 τώρα, κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 76 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε χωριστά για το αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ της παραγράφου 17. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 83 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ίντα 8, κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επτά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ στην αντιλογική σκέψη γάμα. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συ... 10 με 13 Α, μια στιγμή λέει ο κύριο Μίτσελ. Έχει γίνει κάποιο λάθο νομίζω. Στην 8. Στην 8 έγινε κάποιο λάθο. Ότι απορρίφθηκε. Είπατε ενώ εγκρίθηκε. Μπορείτε να λέξετε παρακαλώ τι έγινε με την 8. Εγώ συμφωνώ. Γιατί όχι. Να ελέγξουμε λοιπόν για την αιτιολογική σκέψη 8. Ξεκινάει ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη 10, 10, 15 υπέρ 13 κατάρα εγκρίνεται. Τώρα, αν μπλοκ ψηφίζουμε 10. 10, όχι δεν μπορούμε, αν μπλοκ. Υπέρ τις 10. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Όχι. Καταπίπτουν οι 14, 15 και 16. 17. Τη λέτε 17 με 22. Unblock. Ωραία. Υπέρ. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται 17 με 22. Τώρα 23. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, citations. Πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τρίτη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε Τελική ψηφοφορία επί της τροποποιημένης έκθεσης. Ψηφίστε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεπώς η έκθεση με 26 ψήφους υπέρ, καμία ψήφος κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε πόσο πολύ ε, την ήθελα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και την γραμματεία για την ε, βοήθειά της. Ευχαριστώ, Ινές. Και τώρα συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Μπέρμαν.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 εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία τώρα, αριθμός 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Ελέγχουμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 18. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται.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 25. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 25. Ναι, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 12-12. Ναι, Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία αριθμός 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά,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 Τώρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τροποποιημένη έκθεση του κύριου Μπέρμαν. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 17 ψηφί υπέρ, 10 ψηφί κατά. Συγχαρητήρια. Τώρα ψηφίζουμε την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Αφρικής για το εμπόριο, την ανάπτυξη και την συνεργασία. Υπέρ. Ηλεκτρονικά. Εντάξει. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ομόφωνα εγκρίνεται με 27 ψήφους. Υπέρ. Στη συνέχεια. Ψηφίζουμε την έκθεση και την προφορική ερώτηση όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τελική ψηφοφορία, άρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Υπάρχει όμως η τροπολογία του κύριου Σβένσον. Άρα ψηφίζουμε τροπολογία πρώτα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ε, προφορική ερώτηση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη προφορίες. Εγκρίνεται η προφορική ερώτηση με 18 ψήφους υπέρ, 8 κατά και μία αποχή. Και τώρα διακόπτει ο κύριος Μίτσελ. Σε σχέση με τη δικιά σας έκθεση και την τροπολογία αριθμός 1 του κυρίου Σβένσον, εσείς είπατε ότι απορρίπτεται, αλλά έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται. Μήπως θα μπορούσατε να ελέγξετε. Έτσι, για να δούμε. C'est là. Donc, nous sommes toujours donc, sur, la, sur la question euh, orale, la maman de M. Svensson. Κοιτάξτε, θα επαληθεύσουμε για την τροπολογία του κυρίου Svensson στην έκθεση που μόλις ε, κάναμε πριν, τη δικιά μου. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι ηλεκτρονικά τροπολογία Σβένσον. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και 13 κατά. Εγκρίθηκε. Ο κύριος Ντίβα αυτή. Κύριε Ντίβα, προσέχετε τι κάνετε, λέει ο κύριος Μίτσελ. Euh, Να ξαναψηφίσουμε λοιπόν για την τελική ψηφοφορία με την τροπολογία του κυρίου Σβένσον. Έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την τροπολογία Σβένσον. Ψηφίζουμε τώρα. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία με 19 ψήφους υπέρ, 8 κατά και καμία αποχή. Ensuite, à la question orale. Μετά λοιπόν την προφορική ερώτηση, τροπολογία 1 του κυρίου Μίτσελ. Υπέρ, κατά, αποχές. Ναι, τώρα Εγκρίνεται. Επτά κατά τμήματα ψηφοφορίες, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Second party, qui est pour... Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ναι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η οκτώ καταπίπτει. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέκα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία για την παράγραφο Τροπολογία 11 λέει πρόεδρος. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι υπορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ε, η ψηφοφορία λίγη. Δεκατρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 13, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται. Η 14 καταπίπτει, 15 τώρα. Κατά τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές, εγκρίνονται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 16. από εδώ και πέρα, επειδή έχουμε μόνο μια διαφορά ψήφου κάθε φορά, μια ψήφο διαφορά μάλλον κάθε φορά, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 16 λοιπόν, υπέρ. Έναρξη της ψηφοφορίας. Υπέρ. Εγκρίνεται. 15 προς 12. κατά τμήματα ψηφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεκαοκτώ. Υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. So, yeah, that's what we, that's what we have done. Nous, avons, nous venons de voter l'amendement 18. Μόλις ψηφίσαμε την τροπολογία 18. Le split vote. Le split vote. Φαίνεται να μπορούμε να διεξαγάγουμε κάποιο συμπέρασμα, Πρόεδρε. Εάν το 16 εγκριθεί, αν η 16 εγκριθεί, δεν γίνεται ψηφοφορία κατά τμήματα. Δεν σημαίνει ότι καταπίπτει η επόμενη τροπολογία. <clears throat> 19. Κατά τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Bon. Alors, donc, amendement, euh, aura... Προφορική τροπολογία 2. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 15 προς 12. Η 20 καταπίπτει. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 21. 21. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας Adopté. Adopté. Ναι. Εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Split vote sur recital A. Κατά τμήματα ψηφοφορία για την ε, αιτιολογική σκέψη α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Amendement 2, qui Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κύριε Μίτσελ, με συγχωρείτε, πρόεδρε, αλλά το ΕΛΚ έχει διαφωνία με την προφορική τροπολογία. Πολύ ωραία. Δεν θα να κρίνουμε την προφορική τροπολογία 3. Κατά τμήματα ψηφοφορία για το 3. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Μισό λεπτάκι να βάλω το σκούφο μου, γιατί πραγματικά δεν γίνεται. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 4. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 15-12. Ήταν δύσκολο, ε. ήταν πολύ κοντά η ψηφοφορία το αποτέλεσμα. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την απόφαση όπως τροποποιήθηκε. Το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, toujours. Nous allons reprendre le travail de notre... Συνεχίζουμε μετά από τις ψηφοφορίες με την ημερήσια διάταξη όπου έχουμε την απαλλαγή του κύριου Κρίσπερμαν. Μας... Θα ξανάρθει εδώ φαντάζομαι, δεν τον βλέπω. Θα αλλάξω λοιπόν τη σειρά στην ημερήσια διάταξη με την άδειά σα και θα περάσω στο σημείο 26 που θα το εξετάσουμε πριν από το σημείο 25 επειδή η κυρία Στρίφλερ είναι εδώ και μας έχει ετοιμάσει μία έκθεση, μια που είναι η μόνιμη συγκήτριά μας για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και θα μας μιλήσει λοιπόν για την επίσκεψη στην επαρχία του Νότιου Κίβου. Πήγε εκεί τέλη Νοεμβρίου και θα μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα, τα πορίσματα της αποστολής αυτής. Η κυρία Στρίφλερ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι όντω μόνιμη εκπρόσωπό σα για θέματα ανθρωπιστική βοήθεια και πήγα στο Νότιο Κύβο, στη Λαϊκή Δημοκρατία, τέλη Νοεμβρίου. Πριν συμμετάσχω στη συνεδρίαση με τις χώρες ΑΚΕ. Πήγα λοιπόν επί τόπου, είδα ε, τους καταβλισμούς όπου στρέφουν ε, οι μετανάστες ε, από τον Μπουρούντι κλπ. Πήγα και στο νοσοκομείο στο Κουβού που είναι υπό τον γιατρό Κουάτσι και όπου εκεί υπάρχουν θύματα και βιασμών που καταλαβαίνετε ότι έχουν μεγάλα ψυχολογικά τραύματα αλλά όχι μόνο ψυχολογικά και σωματικά. Επίσης βρέθηκα και με την υπηρεσία ΕΚΟ εκεί, συζητήσαμε για το θέμα της ασφάλειας στην επαρχία. Θέλω να ευχαριστήσω την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και τους εμπειρογνώμων της που είναι εκεί τόπου, στο Κίβο, που βοήθησαν η αποστολή μας να στεφθεί με επιτυχία. Θεωρούμε ότι η περιοχή εκεί είναι ευάλωτη. Η κατάσταση στα ανατολικά του Κονγκό, ιδιαίτερα στο Κίβου, είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δύσκολη και έχει παρατηρηθεί και επιδείνωση στο νότιο Κίβου. Οι στρατιωτικές δράσεις εκεί από το 2009 και μετά δημιουργούν μια συνεχή αστάθεια και έχουν και επιπτώσεις και στην ανθρωπιστική κατάσταση. Μετακινείται ο πληθυσμός, καταστρέφεται ο κοινωνικός ιστός, υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώνεται. Υπάρχουν 800.000 πρόσφυγες μόνο στο Νότιο Κίβο. Έχουν μετατεθεί οι σειράξεις προς την περιοχή αυτή και γι' αυτό έχουμε τόσους πολλούς μετανάστες. Και η κατάσταση δυσκολεύει επίσης και την ανθρωπιστική μας βοήθεια προς τον κόσμο, εκεί που τη χρειάζεται τόσο πολύ. Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε η κινητοποίηση να παραμείνει και η κοινή γνώμη να μην καθησυχάζεται. 50% ήταν η χρηματοδότηση μόνο πέρυσι, ε, δυστυχώς. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μεγάλες επιπτώσεις διότι αυτό κινδυνεύει να συμβεί και με οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα δώσουν λιγότερα χρήματα. Το Βέλγιο, οι κατοχώρε, η Γερμανία, η Σουηδία είναι χώρες που έχουν μειώσει τη χρηματοδότησή του το 2010 και αυτό θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και το 2011. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε αυτό το τμήμα της χώρας. Και όπως έλεγα, οι νέες ζώνες ε, σειράξεων είναι ζώνες τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε εύκολα πρόσβαση. Άρα ούτε υποδομές υπάρχουν, ούτε ασφάλεια υπάρχει στις περιοχές αυτές. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Αυτό λοιπόν παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την προστασία των πολιτών. Οι κανόνες επίσης για την ασφάλεια των ανθρώπων που προσπαθούν να βοηθήσουν εκεί έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί το προσωπικό να έχει πρόσβαση σε αυτέ τι δύσκολε περιοχέ. Άρα η ανθρωπιστική μα βοήθεια εκεί είναι πολύ περιορισμένη. Επιπλέον, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει με τι οποίε συναντήθηκα στο Νότιο Κίβου μα είπαν ότι υπάρχουν νέα προβλήματα στους δρόμους όπου κυκλοφορούν ε, ομάδες που θα έλεγα ότι δεν ε, είναι και πολύ Το σχέδιο που υπάρχει για την λύση των σειράξεων εκεί έχει αποτύχει. Οι στρατιώτες από την κυβέρνηση προσπαθούν να ελέγξουν ε, τις περιοχές που έχουν ορυκτά. Οι πολίτες υφίστανται τεράστια βία και η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Οι γυναίκες και τα κορίτσια υφίστανται καθημερινά τη γενική ατιμορρησία και το στρατιωτικό κλίμα μέσα στο οποίο ζουν. Ο πληθυσμός είναι θύμα και των εκστρατιών ε, καταστολής από τους διάφορους ε, ανυπότακτους και η παραστρατιωτική αλλά και οι στρατιωτικοί είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν ε, την κατάσταση και το κλίμα στην χώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2010 με ψήφισμά του εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση, για την ασφάλεια του πληθυσμού εκεί που χειροτερεύει συνέχεια. Στο νότιο Κίβο, και εδώ θα σας <clears throat> αναφέρω ένα συμβάν για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο πολύ επιδεινώνεται η κατάσταση. Υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ στρατιωτών και ενός κατοίκου και ο στρατιώτης ε, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πολίτη. Οι κάτοικοι σκότωσαν τον στρατιώτη γιατί αντέδρασαν και συνελήφθησαν αυτοί όμως από το στρατό και την 1η Ιανουαρίου οι στρατιώτες ε, έκαναν ε, ε, βίασαν, πήραν την περιουσία, βίασαν τις γυναίκες. Την επομένη οι αρμόδιοι πήγαν και το μόνο που κατάφεραν να κάνουν είναι να διαπιστώσουν την κατάσταση, τίποτα άλλο. Άρα βλέπετε ότι οι πολίτες είναι μονίμως θύματα εκεί. Η κατάστασή τους είναι πάρα πολύ προβληματική, είναι πάντα θύματα της δράσης των στρατιωτών και των παραστρατιωτικών ομάδων. Δεν έχουν καμία προστασία, αντίθετα υφίσταται συνεχώς βιασμούς από όλες τις ένοπλες ε, ομάδες, κυρίως από τους ΦΑΡ, που κυκλοφορούν εκεί και τρομοκρατούν τον πληθυσμό. Μερικές φορές οι πολίτες έχουν φύγει από περιοχές που θεωρούνται ασφαλείς και έχουν πάει σε παραστρατιωτικές περιοχές για να αποφύγουν ακριβώς την βία των ΦΑΡ. Υπάρχουν, υπάρχει λοιπόν τεράστια βία και οι μονάδες που υπήρχαν για να προστατεύσουν από βιασμούς τον πληθυσμό ε, δεν υπάρχουν πια γιατί δεν υπήρξε ηγεσία στο απέ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών εκεί. τεράστιες περιπτώσεις, λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε διασμών. Δεν καλύπτονται έτσι καλλιώς με προστασία όλες οι περιοχές. Η νομιμότητα του Μονίσκου είναι κάτι αμφισβητήσιμο, παρόλο που ηγείται του στρατού του Κονγκό, ο οποίο θεωρείται υπεύθυνο για πάρα πολλού από αυτού του βιασμού. Η ιατρική βοήθεια προσφέρεται από διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει στην περιοχή. Ο συντανισμό όμω μεταξύ του δεν υπάρχει, άρα η αποτελεσματικότητά του είναι πολύ περιορισμένη όπω καταλαβαίνετε. Γενικά μιλώντα λοιπόν το θέμα του συντονισμού είναι ζωτική σημασία. Η στρατιωτική προσέγγιση είναι ανεπαρκή. Δεχόμαστε ότι τελικά ο δεν κατάφερε να προστατεύσει από τους μαζικού παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη χώρα. Η ανθρωπιστική βοήθεια εξαρτάται όμως από το Μονίσκο που όμως δεν καταφέρει να βοηθήσει αρκετά. Η λύση θα μπορούσε να ήταν πολιτική. Χρειάζεται όμως περισσότερο θάρρος από τη διεθνή κοινότητα. Αν δεν αλλάξει τίποτα, τότε οι άνθρωποι που βοηθούν και προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εκεί θα είναι αναγκαίοι για πολύ καιρό ακόμα. Στην Κινσάσα, όταν είχαμε την κοινοβουλευτική συνέλευση, ε, πρέπει να σας πω ότι απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα από όσα άκουσα εκεί. Γιατί τίποτα δεν υπόθηκε απολύτως για τον πολλαπλασιασμό των βιασμών εκεί. <clears throat> Εμεί προτείναμε και ψηφίσαμε πολλά ψηφίσματα. Πρέπει να είμαστε όμω πάρα πολύ προσεκτικοί με τι εξελίξει και να φροντίσουμε να δοθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση. Χαίρομαι για τόσα κάνει η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει ε, την χρηματοδότηση το 2011 για προγράμματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του κόσμου εκεί. Τέλος, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Με κάποιους αδέρφους που ήταν στην Κινσάσα ετοίμασα ε, μία επιστολή στον ε, συμπρόεδρο, ώστε πριν από κάθε γενική συνέλευση που έχουμε ε, μαζί τους, να μας ενημερώνουν λεπτομερώς για την κατάσταση και τη δημοσιονομική, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Και η Επιτροπή βέβαια είναι εδώ και θα μπορέσει και εκείνη να απαντήσει σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό εκεί. Δεν κατάλαβα τι είπατε από αυτού, πρέπει να ομολογήσω. μιλήσατε κάτι, είπατε... Μιλήσατε για την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό. Εγώ νομίζω ότι βοηθάει τον κόσμο, αλλά αυτό που είπατε εσείς εγώ δεν το κατάλαβα. Εσείς είπατε ότι θέλετε να ενισχύσετε τι εκεί. Ξέρουμε ότι τα χρήματα, απαντάει η κυρία Στίφλερ, δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Μίλησα με ένα καθηγητή ιατρικής που είναι στο νοσοκομείο εκεί και είπε ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, διότι τα χρήματα δεν φτάνουν πάντα στον προορισμό τους. Δεν φτάνουν όλα. Και η ΦΙΝΑΠ Κοιτάξτε, σήμερα τη διαχείριση την έχει η Μονίσκου. Θα έπρεπε να αναλάβει τη διαχείριση αυτή ο ΙΕ. Διότι οι άλλοι συμμετέχουν στους διασμούς συχνά, οπότε τι θέλετε. Θα ήθελα πέρα από αυτή τη συνεδρία, να μιλήσουμε για το ΦΙΝΑΠ, του ΙΟ, του ΟΙΕ δηλαδή, που συχνά είχαν εμποϊκοτάρει οι Ηνωμένε Πολιτείε γιατί τους κατηγόρησαν σε σχέση με τις αυλώσεις στην Κίνα. Λάθος όπως, κατά τη γνώμη μου. Κάνανε ό,τι περιμέναμε να κάνουμε. Οπότε πρέπει να δούμε μήπως μπορούμε να πιέσουμε περισσότερο και τους άλλους χρηματοδότες. Euh, Συγγνώμη που άργησα και έλειπα για λίγο και έτσι δεν άκουσα όλα όσα είπατε. Όμως, κάνατε έναν κατάλογο με τους Ευρωπαίους που ήταν εκεί για το τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στην περιοχή. Όπως και να έχει το πράγμα, θα έπρεπε η ΦΙΝΑΠ να ξαναβρει την νομιμότητά της. Διότι τα δώσαμε όλα στο Μονίσκου. Είτε πρόκειται για βίες, ε, αβία, για βιασμούς κλπ. Θα έπρεπε να το ξαναδούμε αυτό. Δηλαδή πάλι ο Ιένα να λάβει τα ενία. Αυτό μου είπανε και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που είναι εκεί ε, παρόντες. Ο κύριος Αντρέα Κόλεμαν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία διορθώνει πρώτος. Κυρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την κυρία Στρίφλερ Ευχαριστούμε για όσα είπατε. Χαρά μας που σας υποδεχτήκαμε εκεί και σας βοηθήσαμε στην αποστολή σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι για το θέμα των βιασμών, ε, το νοσοκομείο εκεί το στηρίζει με ανθρωπιστική βοήθεια από το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε εκεί εδώ και πολύ καιρό και δεν είναι και καινούριο το πρόβλημα, αλλά πράγματι έχουν φτάσει, έχει πάρει διαστάσεις τεράστιες. Το θέμα όμως των βιασμών δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο και έχει να κάνει με την προστασία των πολιτών. Γιατί γίνονται και άλλα. Γίνονται συλλήψεις που δεν θα έπρεπε. Υπάρχει ατιμορρησία, γενικευμένη. Ε, μαζεύουν παιδιά και τα κάνουν στρατιώτες. Άρα τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να απομονώσουμε τους βιασμούς από τα υπόλοιπα, διότι έτσι στιγματίζουμε, αν μου επιτρέπετε να το πω, και γίνεται και λίγο σεξι, έτσι, ελκυστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Θα έπρεπε να δώσουμε την ίδια προσοχή σε όλες τις πτυχές του προβλήματος αυτού. Η ανθρωπιστική βοήθεια ανακουφίζει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Η απάντηση όμως θα έπρεπε να είναι διαρθρωτική, δηλαδή να μην υπάρχει ατιμορρησία, να υπάρχει το κράτος στις περιοχές αυτές κλπ. Τώρα η Μανούσκο συντονίζει την κατάσταση όσον αφορά τους βιασμούς και ο ΙΕ συλλέγει δεδομένα. Αυτό κάνει. Που είναι και αυτό σημαντικό πολύ. Όντως, ο συντονισμός είναι λυπής. φτιάξαμε ε, ένα κλάστερ προστασίας, κάτω από το οποίο προσπαθούμε να υπάρχει συντονισμός. Στις ανατολικές επαρχίες υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν ξεκινήσει να οργανώνουν έναν άτυπο συντονισμό. Πράγματι πρέπει να υπάρχει ο συντονισμός, γιατί Μόνο έτσι η Μονισκό θα μπορέσει να παίξει πραγματικά το ρόλο της. Αναφέρατε επίσης και την ε, μη πρόσβαση σε διάφορες περιοχές. Τόσο στο Κίβο όσο και στις ανατολικές επαρχίες υπάρχει το Lord Resistance Army. Πάνε στις πιο απομονωμένες περιοχές και ζουν με τον πληθυσμό. Και όταν πάνε ένοπλες δυνάμεις για να παρέμβουν, τα βάζουν και αυτοί με τον πληθυσμό. Οπότε είναι διπλά θύμα ο πληθυσμός εκεί. Πρέπει σίγουρα να υπάρχει συνεργασία και να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στις υποδομές. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και με το νοσοκομείο πάντως δουλεύουμε για να υπάρχουν ε, μονάδες που μετακινούνται. Και υπάρχει μια στρατηγική ενίσχυση της δυνατότητας που έχουν τα κέντρα υγείας του Κονγκό για να αντιμετωπίσουν ε, βιασμούς μέσα στις πρώτες ώρες. Και έχουμε και στήριξη μέσω της EcoFlight, που είναι μια υπηρεσία πτήσεων που επιτρέπει στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να πηγαίνουν στις πιο απομονωμένες περιοχές και να βοηθούν όσο γίνεται περισσότερο. Πρόεδρος, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 23, 24 και 25 που έχουν να κάνουν με τις απαλλαγές. Ο κύριος Μπέρμαν έχει ετοιμάσει δύο γνωμοδοτήσεις και ο κύριος Γκέρενς έχει μια τρίτη γνωμοδότηση για την απαλλαγή. Έχουμε δύο εκθέσεις του Λεγκτικού Συνεδρίου που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΦΕΔ στην περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση της Ανατολικής και Δυτικής Αφρικής. Θα εξετάσουμε τις τρεις αυτές γνωμοδοτήσεις μαζί. Κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις γνωμοδοτήσεις ερωτήσεις σας. Και τις δύο μαζί, έτσι λέει ο κύριος Μπέρμαν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Στα Ολλανδικά. Οι δύο αυτές γνωμοδοτήσεις έχουν πολλά κοινά, αλλά θα ξεκινήσω με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αυτό που είναι ξεκάθαρο και είναι θετικό είναι ότι μιλάμε για την ακρίβεια όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο. Καλός έλεγχος λοιπόν που μας γίνεται απ' έξω. Ωραία. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό είναι η βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού στις διάφορες αντιπροσωπείες. Και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν ε, οι διαδικασίες προσφορών, υπάρχει ο έλεγχος που γίνεται από τις αντιπροσωπείες και υπάρχει και ο εσωτερικός έλεγχος. Και για τα τρία αυτά, και εξάντε και εσωτερικός έλεγχος και προσφορές, πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ό,τι ελλείψεις παρατηρούνται εκεί και αδυναμίες. Παρατηρεί το ελεκτικό συνέδριο ότι λείπει η δημοσιονομική στήριξη. Δεν μας εκπλήσει αυτό, πρέπει να πω. Πάντως, οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τις ακολουθήσουμε. Να δούμε τις μεθόδους μας για την επαλήθευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πιο συγκεκριμένα να προσπαθεί να ε, βρίσκει τους ελέγχους και τους ε, μετά ελέγχους που γίνονται. Για να μην υπάρχει αυτό το αδύναμο σημείο που συζητιέται και στα Εθνικά Κοινοβούλια. όσον αφορά τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Τέλος, τις αντιπροσωπίες στις διάφορες χώρες υπάρχουν ελλείψεις στο προσωπικό, πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότητα του έργου μειώνεται και είναι κρίμα. Τώρα, για την άλλη γνωμοδότηση σχετικά με το γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ διαπιστώνονται λιγότερα λάθη και λήψη από ό,τι κατά το παρελθόν. Πάντως, η ΕΚΟ θα μπορούσε να έχει καλύτερο έλεγχο. Το κοινοβούλιο, οι κοινωνίες, ε, τα κοινοβούλια μάλλον, οι κοινωνίες των πολιτών θα μπορούσαν να αναμειχθούν περισσότερο με μια κατάλληλη στρατηγική και να παίξουν ένα πιο σημαντικό ακόμα ρόλο. Η κοινωνία των πολιτών λοιπόν και τα εθνικά κοινοβούλια. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε, να γίνεται μεγαλύτερος και να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στις διάφορες χώρες. Δυστυχώς ούτε αρκετά χρήματα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είπαμε λήψεις και στο προσωπικό και στον προϋπολογισμό. Τέλος, 20% του προπολογισμού έχουμε πει ότι θα πηγαίνει στην υγεία και στην εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιμείνει στην απέτηση αυτή. Είναι αναγκαίο και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δείξει με ποιο τρόπο, με τι μέσα θα προσπαθήσει να πετύχει, ώστε η απέτηση αυτή που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό θα τηρείται. Ιδιαίτερα για την υγεία υπέρ των γυναικών. Η θνησιμότητα στη γέννα παιδιών και μητέρων δυστυχώς εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να βελτιωθεί. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα σχολιάσω την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 18 του 2009 για την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη και της περιφερειακής ολοκλήρωσης στην ε, Ανατολική και Δυτική Αφρική. Εδώ θέλω να κάνω το εξή σχόλιο. Εδώ βλέπουμε ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση ε, δημιουργεί θέσεις εργασίας και απασχόληση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Και στην έκθεση αυτή εκφράζουμε την ικανοποίησή μα για το ότι οι χρηματοδοτήσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη συνοδεύτηκαν το 2009, μάλλον διπλασιάστηκαν το 2009. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει στην Αφρικανική Ήπειρο είναι η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο για πολλαπλού λόγου. Τα αφρικανικά πρότυπα πολύ συχνά αντιγράφονται με βάση τα ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως επιτελείται ταχύτερη πρόοδος όταν υπάρχει συνεργασία περιφερειακή. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως ε, για την ε, Δυτική Αφρική. Και βέβαια ακόμη η χρήση των κοντιλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Αυτό για διαφορετικούς λόγους Το βλέπει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χειρίζεται το εν λόγω ταμείο. Όμω η ικανότητα απορρόφησης ε, των ε, κονδυλίων αυτό από την πλευρά των Αφρικανών, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, δυστυχώς δεν είναι επαρκή Η περιφερειακή διάσταση για την ώρα χρήση στήριξη ε, για σκοπούς ανάπτυξιακή βοήθειας. Βέβαια βλέπουμε να έχει γίνει πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Και σε κάθε περίπτωση η περιφερειακή συνεργασία δεν είναι κάτι το απλό επειδή επικαλύπτονται πολύ διαφορετικοί οργανισμοί εδώ. Τα πράγματα είναι εξίσου πολύπλοκα όπως και στην Ευρώπη φαίνεται. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι μέλη μιας οργάνωσης και ταυτόχρονα μιας άλλης, όπως η Σενεγάλη που είναι μέλος της ε, Νομισματικής και ε, Οικονομικής Ένωσης της, Δυτικό, της Δυτικής Αφρικής, αλλά και της ΕΝΤΕΑΟ, δηλαδή Υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξία, αλλά υπάρχουν και κάποιε δυσκολίε. Υπάρχουν και οι συμφωνίε οικονομική συνεργασία, περιφερειακή εμβέλεια, που όμω δεν έχουν παντότε την ίδια κάλυψη με τι ευρύτερε οργανώσει ε, τη γεωγραφική αυτή περιοχή. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να μας πληροφορήσει αν θεωρεί ότι ε, στηρίζονται παρκώ όλε αυτέ τις προσπάθειε. Εγώ δεν είμαι σε θέση να εκφράσω την ε, τελική μου άποψη και θα προτιμούσα να ακούσω πρώτα και την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σημαντικός δωρητής σε αυτήν την περιοχή, ιδίω στο capacity building, στην οικοδόμηση δυνατοτήτων, μπορεί να προσφέρει τα περισσότερα για να απεμπλέξει κάποιες περίπλοκες περιφερειακές καταστάσεις και να αποφευθούν και οι επικαλύψεις. Η αφρικανική οικοδόμηση σε περιφερειακό επίπεδο είναι ε, οικοδόμηση για όλη την Ήπειρο. Οφελεί όλους τους Αφρικανούς. Μπορούμε να συνοδεύσουμε λοιπόν αυτήν την ε, τάση που υπάρχει, να προσφέρουμε την πείρα μας και τις εμπειρίες μας ε, προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι. Και έπειτα συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό θα ήταν να μην ασκήσουμε υπέρματρη πίεση ε, στους τοπικούς πληθυσμούς για την υπογραφή οικονομικών, ε, συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας και οικονομικής εταιρικής σχέσης. Όμως ε, η περιφερειακή συνεργασία που επιθυμούμε θα υποβοηθεί το ιδιαίτερα από κάτι τέτοιο. Τώρα, για την ειδική έκθεση 15 του 2009 που αφορεί, αφορά την κοινοτική συνδρομή για τη στήριξη του ΟΗΕ. Εδώ καλό θα ήταν να, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ευνοϊκό για τις οικονομίες κλίμακας με όλα τα δυνατά μέσα και μέσω του ΟΗΕ να φτάσουμε σε περικοπή του κόστους, ιδίως σε συγκεκριμένους τομείς. Όμως θα ήταν αυταπάτη να υπολογίζουμε μόνο στους μεγάλους θεσμικούς φορείς. Ξεχνάμε την κοινωνία των πολιτών που είναι πολύ σημαντική για την ιδιοποίηση των προγραμμάτων. Εάν δεν αναλάβουν ίδια την ευθύνη των προγραμμάτων αυτών, χάνουμε μια από τις βασικές αρχές, μια από τις θεμελιώδεις αρχές κάθε περιφερειακής ανάπτυξης και τεχνικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να είναι όσο για δυνατόν πιο διαφανή και πιο δραστική, ώστε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα τη βοήθεια. Δεν θέλω να είμαι ιδιαίτερα επικριτικό κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα και να την ακούσω. Τα σχόλιά τη, ιδίω σε σχέση με όσα παρατήρησε το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτά λίγο πολύ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Και λυπάμαι που η παρέμβασή μου, όπως είπε και ο φίλος Τάις, έγινε ε, εν πλήρη κοινοβουλευτική αδιαφορία. Το λόγο έχουν οι υπόλοιποι βουλευτές που θέλουν να τοποθετηθούν. Όχι, κανεί δεν θέλει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπέλινγκτον. Με συγχωρείτε. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι θα ευγνώμονες για τα σχόλια των δύο εισηγητών για τα δύο θέματα. Θα προσυπογράψω αυτό που είπε ο κύριος Μπέρμαν για τη γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το EDF. Μετά από κάποια χρόνια μπόρεσε να πει το συνέδριο ότι η διαχείριση του Ταμείου δεν επηρεάζεται από ουσιαστικό σφάλμα το 2009 και αυτό μας ενθαρρύνει πολύ. Επίσης σημειώσαμε ότι το ποσοστό των συναλλαγών που επηρεάζεται από σφάλμα μειώνεται διαχρονικά από το 2007 και μέχρι το 2009. Η μείωση είναι στατιστικά σημαντική. Οπότε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πιστεύουμε ότι άρχισαν πια να δίνουν καρπούς εις ό,τι αφορά τον έλεγχο από το συνέδριο. Επίσης μας ενδιαφέρει να επιτελέσουμε περαιτέρω πρόοδο. Επίτροπος Πίμπολ ξανακοίνωσε στην ακρόαση στην Επιτροπή Κοκομπίου στις 13 ε, Ιανουαρίου ότι είναι αποφασισμένος να κάνει μια ανασκόπηση, αναθεώρηση της ελεγκτικής πυραμίδας των συστημάτων ελέγχου ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι αποτελεσματικά και αποδοτικά για τον έλεγχο των δαπανών. Ξέρουμε ότι δουλεύουμε σε... Ε, ε, περιοχή ψηλού ρίσκου εις ό,τι αφορά τα καταπιστεύματα. Επίσης ε, έχουμε και κάποιον οδηγό που βοηθεί τον καλύτερο έλεγχο από τις αντιπροσωπείες και έχουμε και ένα toolkit σαν με σειρά εργαλείων για τις ε, υπεύθυνες μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την υλοποίηση, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν, να ακολουθούν τους κανόνες μας αυστηρά και να γίνεται καλύτερη εφαρμογή ε, σύμφωνα με τους κανόνες. Τώρα, για την δημοσιονομική στήριξη. Όπως είπε ο κ. Μπέρμαν, αληθεύει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο παρατυπιών που εντοπίστηκαν από το Ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά τις ε, επιχειρήσεις με δημοσιονομική στήριξη. Οι περισσότερες ήταν τυπικές, χωρίς δημοσιονομικό αντίκτυπο και υπάρχει σημαντική βελτίωση μετά από την εισαγωγή του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και στις δημοσιονομικές συμφωνίες για το 10ο EDF και τις, ε, οι επιχειρήσεις δημοσιονομικής στήριξης τροποποιήθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στα μελήματα του ελεγκτικού συνεδρίου και έτσι επετελέστη σημαντική πρόοδος, βελτίωση. Για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις ελεγκτικές ικανότητες συμμεριζόμεθα εν πολύ στην ανησυχία του Κοινοβουλίου εδώ και το ότι τα κοινοβούλια τα εθνικά σε μια χώρα εταίρο θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των δαπανών. Αυτό πάντα το λέγαμε για τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, δηλαδή τα συστήματα τοπικής παρακολούθησης και ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται και εμείς εργαστήκαμε με το Κοινοβούλιο και μπορούμε από κοινού να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα για τη βελτίωση αυτών των ε, δράσεων. Μόλις φύγω από εδώ θα πάω σε μια συζήτηση που οργανώθηκε από το OPPD σας με βουλευτές από την Κεντρική Αφρική. Είναι σημαντικό λοιπόν να προωθηθεί ο διάλογος αυτός, να ενθαρρυνθεί. Τώρα, για τις προσλήψεις, το προσωπικό των αντιπροσωπιών, ο Επίτροπος Πίμπαλ ξανακοίνωσε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών ότι προτιθέμεθα να προετοιμάσουμε μια στρατηγική μακροπρόθεσμη για το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να συμπαντίζει το προσωπικό με τους μακροπρόθεσμους στόχους και με την δημιουργία της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης η ευθύνη για το προσωπικό που εργάζεται σε αντιπροσωπείες για την αναπτυξιακή βοήθεια πέρασε από την παλιά Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΚ στη νέα, την Γενική Διεύθυνση ΝΤΕΒΚΟ. Οπότε υπάρχει τώρα πολύ πιο στενή σχέση με το προσωπικό που εργάζεται σε αντιπροσωπείες πάνω σε αυτά τα θέματα και θέλουμε να βελτιώσουμε και το συντονισμό σε αυτό το τομέα. Για το όριο το συγκριτικής αξιολόγησης, ας πούμε 20%, χαίρομαι μπορώ να σας πω ότι το ποσοστό που μου δώσανε για το 2009 ήταν 22,6% στη DCI, το μέσο ανεπτυξιακής συνεργασίας, δηλαδή φτάσαμε στο μέτρο συγκριτικής αξιολόγησης το 2009, το benchmark, και οι εκτιμήσεις για το 2010 μας πάνε στο 23,2% με μια μικρή αύξηση δηλαδή, οπότε συμφωνούμε και με τους στόχους που έχουν τεθεί σε αυτό το τομέα. Όταν δεχτήκαμε, συμφωνήσαμε για το benchmark στις διαπραγματεύσεις για το DCI, είμαστε ε, πεπισμένοι ότι θα έπρεπε μέχρι το, την ενδιάμεση αξιολόγηση να είχαμε φτάσει στο στόχο αυτό. Και αυτό έγινε. Τώρα θα προσπαθήσω να συντομεύω για να δούμε τώρα το θέμα της ορατότητας που έθεσε ο κύριος Μπέρμαν στις προτάσεις του για τις εκθέσεις απαλλαγής. Δουλέψαμε στενά με τα Ηνωμένα Έθνη για την ορατότητα. Συμφωνούμε συμφωνήσαμε για κατευθυντήριες γραμμές ε, κοινέ για την ορατότητα πριν από λίγες χρόνια. Ε, υπήρχε και ένας εκπρόσωπος από τη UNWA ε, που κουβαλούσε μια τσάντα που είχε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λογότυπο ακριβώς σύμφωνα με τις κατευθυντηρίες γραμμές για την ορατότητα. Οπότε είδα τα μάτια μου την ε, βελτίωση και την πρόοδο εκεί. Τώρα για το θέμα, τα θέματα του κυρίου Γκέρντς, για την ε, περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση καταρχήν Δουλέψαμε σκληρά για να επιτελέσουμε πρόοδο στο ποσοστά απορρόφησης που αποτελούν ακόμη πρόβλημα. Εγώ έτρεξα το πρόγραμμα για την ε, Ανατολική Αφρική ο ίδιος και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να συνεχίσει η εξέλιξη. Πάντως ε, έχουμε εκτιμήσει ότι για την Ανατολική και Νότια Αφρική, θα χρησι... Ε, τη Μεσημβρινή Αφρική, θα χρησιμοποιηθούν σίγουρα μέχρι το 2013 τα διαθέσιμα κονδύλια. Οπότε και εδώ έχουμε πρόοδο. Τώρα για τη Δυτική Αφρική δεν μπορούμε ακόμα να δώσουμε ημερομηνίες, αλλά δουλέψαμε σκληρά και στους δύο τομείς για να βελτιώσουμε τη συνοχή μεταξύ περιφερειακής και εθνικής στρατηγικής. Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες συστάσεις από τις εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τον Οκτώβριο του 2010 εκδώσαμε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για όλο μας το προσωπικό για τη διαχείριση των περιφερειακών προγραμμάτων και ειδικότερα εξετάσαμε το θέμα που έθεσε το ελεκτικό συνουνέδριο που δεν κατέληξε σχετικά με την αποτελεσματικότητα και υπάρχει μια εξατομικευμένη αξιολόγηση. Πάλι θα συνεργαστούμε με το, τα Ηνωμένα Έθνη εκ του σύνεγγης, γιατί έχουμε κοινέ ε, προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων και τις δράσεις παρακολούθησης των δικτών εισρώων νεκρών. Ε, ε, πρόσφατα συμφωνήσαμε για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εκθέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη και το 2009 τον Ιούνιο εκδώσαμε οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες μας λέγοντας ότι χρειάζεται σαφέστερη τεκμηρίωση τυχόν προτάσεων για να περάσουν κονδύλια από το Ηνωμένα Έθνη ή τις διεθνείς οργανώσεις. Θα έπρεπε δηλαδή να εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία πριν χρησιμοποιηθούν αυτοί οι διάβλοι. Οπότε ελπίζουμε ότι αυτό θα ανταποκρίνεται και θα καλύψει την σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου μέσα από τη δράση αυτή με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο κύριος Μπέρμαν. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι χρειάζεται συζήτηση εις βάθος ε, σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς αξιολογεί η ίδια τους κανόνες αυτούς, 20% τουλάχιστον για τον υγειονομικό τομέα και την εκπαίδευση και ποια είναι τα ωφέλη, τα πλεονεκτήματα και ενδεχομένως και τα μειονεκτήματα. Πρέπει να το συζητήσουμε εις βάθος. Κατά δεύτερο, δεν θα συμφωνήσω με τις φωνές όσων ομαδικά κατακρίνουν την, τον ΟΗΕ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια στρατηγική η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιδιώκει μια δική της στρατηγική για να ενισχύσει την αναπτυξιακή βοήθεια από μόνη της. Υπάρχουν, ε, υπάρχει ο ΙΕ γι' αυτό και θα πρέπει να επιδιώξουμε την ε, προώθηση των, ε, της δικής μας βοήθειας μέσω του ΟΗΕ. Θα ήταν στρατηγικό σφάλμα να επιδιώξουμε κάτι τέτοιο. Ο ΟΗΕ βρίσκεται παντού. πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους διάβλους που μας προσφέρει. Και είναι πολύ εύκολο να το κατακρίνουμε και γι' αυτό. Επίση υπάρχουν διαφορέ ε, λογιστικέ μεταξύ ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δεν είναι επαρκή λόγο για να μην ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάβλο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών σήμερα, 27, την 5η μάλλον, 27 Ιανουαρίου, το μεσημέρι θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μα έκθεση τον Φεβρουάριο. Ε, κλείνουμε με αυτό το θέμα και περνάμε στην αποστολή στο Νεπάλ παρουσίαση από τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας της ΔΕΒΕ, κύριο Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ έφερε πέρας με μεγάλη επιτυχία την αποστολή αναπτυξιακή στο Νεπάλ στις 27 Σεπτεμβρίου και χάρη στη συνεργασία των κυρίων Ντέβα, Λαμπέρ, Ρινάλντι, της κυρίας Μάιλον Λαμπέρ, επικεφαλής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις συνεργασίας με τις χώρες της Νοτιού Ασίας, όλα πήγαν καλά. Το έγγραφο που έχετε στο φάκελό σα ολοκληρώθηκε στο τέλο του 2010. Ακόμη και αν ο κ. Γκερέρο δεν μπόρεσε να έρθει τον Δεκέμβριο εξαιτία του πρόσφατου διορισμού του ως επικεφαλής της ομάδας ε, για τα συνταγματικά θέματα στην πολιτική του ομάδα, όμως θα συνεχίσει να συνεισφέρει στο δικό μας έργο, έστω και από εκείνη τη θέση και χωρίς να καθυστερήσω περαιτέρω, θα του δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει τα βασικότερα σημεία από την αποστολή αυτή. Κύριε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Οι λίγοι που έχουν μείνει εδώ θέλω να παραμείνουν φίλοι μου, μην τους χάσω. Οπότε θα είμαι σύντομος. Όπως λέγαμε, ήμασταν ο κύριος Ντέβα, ο πρόεδρος, ο κύριος Ρινάλντι από τους Φιλελεύθερους, Ιταλία, η κυρία Λάμπερτ, η οποία είχε πάει και νωρίτερα στο Νεπάλ, πρόεδρος μιας αντιπροσωπείας για την Ασία πιο πολιτικού χαρακτήρα. Και ήμουν και εγώ πρόεδρος της αντιπροσωπείας αυτής. Στόχος μας κυρίως ήταν να ελέγξουμε πώς λειτουργούν τα θέματα ανάπτυξης στο Νεπάλ. Ιδιαίτερα τι έχει να κάνει με τη χρηστή διακυβέρνηση. Κάτι πολύ σημαντικό σε μια χώρα που πέρασε εμφύλιο για χρόνια και τώρα είναι στη διαδικασία ανοικοδόμησης και ειρήνευσης. Και όσον αφορά το περιβάλλον, η χώρα πλήττεται από τις κλιματικές αλλαγές. Συχνά υπάρχουν ε, κίνδυνοι πλημμυρών. Ένα άλλο θέμα ήταν η εκπαίδευση, γιατί ακριβώς εξαιτία του εμφυλίου πολέμου η χώρα για χρόνια αναγκάστηκε να κρατήσει τα παιδιά μακριά από τα σχολεία. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλά μέλη της κυβέρνησης του Νεπόλ και Υπουργό Εξωτερικών και Εκπαίδευσης, Ανοικοδόμησης, με εκπροσώπους επίσης της ε, Ιδρυτικής Συνέλευσης που είναι πολύ σημαντική γιατί ακριβώς ετοιμάζουν ένα νέο σύνταγμα. Όπως επίσης συναντηθήκαμε και με την Εκλογική Επιτροπή που και αυτή είναι σημαντική διότι στο εγγύς μέλλον θα λάβουν χώρα εκεί εκλογές και η Επιτροπή αυτή έχει ε, μεγάλη πολιτική σημασία. Δεν συναντηθήκαμε όμως μόνο με επίσημα όργανα, συναντηθήκαμε και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είχαμε μια διακριτική συνάντηση με μια οργάνωση γυναικών που αγωνίζονται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους ενός Διεθνούς Κέντρου ε, Ανάπτυξης ε, της Υπέθρου σε ορεινές περιοχές. Ε, επισκεφθήκαμε ένα δημόσιο σχολείο και επισκεφθήκαμε και ένα κέντρο που διαχειρίζονται γυναίκες από τους Δαλίτ, που είναι μια μειονότητα εκεί. Η κατάσταση στο Νεπάλ, τα λέει και η έκθεση, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, είναι η εξή. Το Νεπάλ πέρασε από μια μακρά περίοδο εμφυλίου πολέμου και τώρα προσπαθεί να πετύχει την ειρήνη και την ανοικοδόμηση. Ετοιμάζει και ένα νέο σύνταγμα έχει μια κυβέρνηση η οποία εκτελεί ε, χρέη κυβέρνηση, χωρί όμω να έχουν γίνει εκλογέ και να έχει εκλεγεί ένα πρωθυπουργό. Υπάρχει πρόοδο σύμφωνα με τον δίκτυο ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά έτσι κι αλλιώ η χώρα βρίσκεται πίσω γιατί είναι στην 136η θέση από τις 180 χώρες που περιλαμβάνει ο κατάλογος. Μιλήσαμε για τη διευκόλυνση του διαλόγου και θέλουμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και γείτονες του Νεπάλ. Από πάνω το Θιβέτ και η Κίνα και από κάτω η Ινδία είναι χώρες που τους ενδιαφέρει να αναλάβουν ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή, να έχουν εκείνες το πάνω χέρι. Οπότε, στο Νεπάλ πρέπει να υπάρχει μια τρίτη λύση μια συνένεση για λύσεις όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα όσον αφορά την αναπτυξιακή μας πολιτική. Και εδώ πρέπει επίσης να σημειώσω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Ιανουαρίου κατέληξε σε μια συμφωνία με τον ΕΠΑΛ και κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης για μια συμφωνία πολιετή 2011-2013 είναι κάτι θετικό και το στηρίζουμε. Το μεγαλύτερο μέρος, 60 εκατομμύρια, είναι εκπαίδευση, ειρήνη, πολιτική σταθερότητα, εμπόριο και οικονομική ανάπτυξη. Αυτοί είναι οι κύριοι τομείς που περιλαμβάνονται στο Country Strategy Paper. Τα 60 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αύξηση κατά 33% της δικιάς μας αναπτυξιακής συνεργασίας με τον ΕΠΑΛ. Καλό είναι αυτό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η αντιπροσωπεία μας με ικανοποίηση διαπίστωσε την πρόοδο που επετέχθη με το μνημόνιο αυτό, το υπογραμμίζουμε και τώρα, και θεωρούμε ότι αν συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία στον ΕΠΑΛ, αν συνεχίσουμε την πρόοδο στην εκπαίδευση, το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη και αν συντονίσουμε καλύτερα την προσφορά των δωρητών, θα μπορέσει και τον Νεπάλ να πετύχει τους στόχους της χιλιετίας το 2015. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας που με συνόδευσαν στο ταξίδι αυτό. Τον Ραφαέλε, την Πέτρα, την Ελένα Μουνιώθ επίσης, που βοήθησε να γίνει το ταξίδι αυτό και καρποφόρο αλλά και να έχουμε την παρουσίαση που σας προσέφερα μόλις τώρα. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχουν τώρα οι βουλευτές. Ο κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για τον Ερικέ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο Νεπάλ, μπορέσετε να μιλήσετε για το μέσο διευκόλυνσης για τα τρόφιμα. Το ένα δις για να προωθηθεί η αγροτική ανάπτυξη σε πολλές αντισώμενες χώρες εκ των οποίων το Νεπάλ. Έχετε νέα για το τι συνέβη με αυτό το κονδύλι. Όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γεωργία και συγκεκριμένα όσον αφορά τη στήριξη στους αγρότες, τους τοπικούς εκεί, τι καλλιέργειες μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις στις κλιματικές αλλαγές, δεδομένων των παγετών στο Νεπάλ, όλα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο προηγούμενης επίσκεψης από το Κοινοβούλιο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την περιοχή, της οποίας πρόεδρος είναι η κυρία Λάμπερτ. Οπότε, εμείς είχαμε ως στόχο στην επίσκεψή μας να δούμε μεν και τις δυσκολίες με τη Γεωργία, αλλά αυτές αναλύθηκαν περισσότερο από την προηγούμενη αποστολή που πήγε εκεί το Μάιο του 2010, δηλαδή μόνο πέντε μήνες πριν πάμε εμείς. Τα προβλήματα πάντως της γεωργίας επισητιστικής ασφάλειας στο Νεπάλ και δυνατότητες βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν αντικείμενο των συζητήσεών μας. Γιατί, όπως σας είπα, οι κλιματικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τον Νεπάλ και η κατάσταση είναι πολύ λεπτή λόγω της γεωγραφικής θέσης του Νεπάλ. Ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ και συγχαίρω τον συνάδελφο κύριο Σάλμον για την πολύ καλή διεξαγωγή της αντιπροσωπείας. Μάθαμε πολλά. Έχω πάει πολλές φορές στο Νεπάλ και ανησυχώ διότι ακόμη δεν μπορούν να σχηματίσουν σωστή κυβέρνηση. 18 φορές έχουν αποπειραθεί. 18 φορές. Τα τεκτενόμενα στο Βέλγιο φαίνονται παιδιάστικα πράγματα και δεν τα καταφέρνουν. Εκτός αυτού μου λένε τώρα ότι τα Ηνωμένα Έθνη ε, σχεδιάζουν να αποχωρήσουν Υπάρχει ο στρατός, οι Μόροι που έχουν αφοπλιστεί και τα Ηνωμένα Έθνη που ε, ήταν, αν θέλετε, ένα σταθεροποιητικό φράγμα, το οποίο τώρα αποχωρεί και δεν υπάρχει και κυβέρνηση στη χώρα θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποια μόχλευση εκεί. Είμαστε άλλωστε από τους ε, μεγαλύτερους δωρητές. Μας ενδιαφέρει η χώρα. Ε, είναι ε, πάνω στην σεισμική ζώνη των Ιμαλαίων. Είναι πολύ έντονο το λιώσιμο των παγετώνων και μπορεί να υπάρξουν πλημμύρες ε, λόγω των λιμνών, ε, των λεκάνων, λεκανών ε, συλλογής υδάτων κλπ. Και όλα αυτά γίνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Επίσης έχουμε τις πλημμύρες στο Πακιστάν πάλι λόγω της κλιματικής αλλαγής και το Νεπάλ είναι πολύ εύθραυστη χώρα έχει μια δομική, κατασκευαστική ε, ε, αδυναμία. Τα κτίρια δεν αντέχουν. Υπάρχουν τα θέματα των τροφίμων, της σταθερότητας, ε, πολλά προβλήματα συσσωρεύονται και πολλές ανάγκες πρέπει να αντιμετωπιστούν, πολλά να διορθωθούν γρήγορα άκουσα γιατί μίλησα σε έναν φίλο εκεί πριν από λίγες μέρες ότι κόβεται το ρεύμα για 16 ώρες ε, ενώ υπάρχει ε, μεγάλο ηλεκτροπαραγωγό δυναμικό από τα νερά που κατεβαίνουν και δεν γίνεται τίποτε και μένει η χώρα στο σκοτάδι από τις διακοπές του ρεύματος. Πρέπει λοιπόν κάποιος να τα θέσει αυτά υπό έλεγχο. Οι ίδιοι κάτοικοι του Νεπάλ δεν κατάφεραν να τα καταφέρουν οι ίδιοι. Αυτό που θέλω να πω είναι να γίνει ίσως μια περιφερειακή διάσκεψη με μας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα δράσει διευκολυντικά, για να δούμε πώς θα βοηθήσουμε. γιατί θα πρέπει και οι χώρες γύρω από τον Νεπάλ να βοηθήσουν, να συνδράμουν τους κατοίκους του Νεπάλ που είναι σε τόσο δύσκολη θέση. Οι διμερείς μας σχέσεις με το Νεπάλ είναι εξαιρετικές. Και λοιπόν όμως τους δίνουμε υποστήριξη και χρήματα όποτε μπορούμε, αλλά δεν βελτιώνουμε τις προοπτικές τους έτσι. Σκέφτομαι δυνατά λοιπόν και λέω ότι ίσως θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε μια περιφερειακή διάσκεψη με χώρες της περιοχής, με μας, με άλλους δωρητές ενδεχομένως, τις Ηνωμένε Πολιτείε που βοηθούν και αυτές και τέλος πάντων όποιον άλλον θέλει να έρθει και να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι με όλους τους προθύμους και τους ε, ε και να δούμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα με μια σειρά από θέματα. Αλλιώς όλα είναι στον αέρα. Και η ε, βοήθειά μας έτσι δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι αποτελεσματική. Έχετε δίκιο, πολύ καλή πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Κανεί δεν είναι εδώ από την Επιτροπή. Να δώσω λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο Γκερέρο για να ολοκληρώσει αν θέλει. Ναι, απλώ να επισημάνω ότι την περασμένη εβδομάδα ή πιο σωστά πριν από 12 ημέρες η πιο σωστα πριν απο 12 ημέρε η αποστολη του ΟΗΕ στο Νεπάλ ολοκληρώθηκε ε, και έφυγε, έφυγαν οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ από το Νεπάλ. Υπάρχουν ακόμη ανησυχίες για την ένταξη των μαοϊστών στο στρατό του Νεπάλ, το κατά πόσο θα έχουν πια όπλα στα χέρια τους και ούτω καθεξής. Πάντως το θετικό νέο είναι ότι την επόμενη μέρα από την αναχώρηση του ΟΗΕ, οι Μαοϊστές υπέγραψαν μια συμφωνία όπου δεσμεύονται εκ νέου να συμμετάσχουν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Υπάρχει λοιπόν μια βελτίωση σε σχέση με όσα αναμένονταν μετά την, περίοδο μετά την αναχώρηση του ΟΗΕ. Βεβαίως, Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που ανέφερε και ο συνάδελφος ε, Ντέβα στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και στι μελλοντικέ μα συζητήσει στην Επιτροπή. Και σίγουρα η περιοχή αυτή επηρεάζεται από τι κλιματικέ αλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παράγουμε περισσότερη ενέργεια, να μπορεί η χώρα αυτή να είναι αυτάρκη και να βελτιώσουμε την κατάστασή τη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, μειονότητα τάρι που επισκεφθήκαμε, είδαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί παράγουν γεωργικά προϊόντα και πειραματίζονται με νέα προϊόντα εκεί. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα στο πρωτόκολλο Συμφωνία Συνεργασίας Αλληλευτικής μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Μικρονησίας. Συζήτηση για αλληλευτική συμφωνία και πάλι. Εδώ θα τοποθετηθεί η Επιτροπή μα ό,τι αφορά την αλληλευτική αυτή συνεργασία, εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μικρονησία. Κύριε Ντέβα, είστε συγκεκριτή μα για αυτή την ε, γνωμοδότηση. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι αλληλευτική συμφωνία που έληξε στις 21 Φεβρουαρίου και θέλουμε να την παρατείνουμε με τη διαδικασία συγκατάθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Είμαστε πρόσφατα στην ε, περιοχή όταν εξετάσαμε τις συμφωνίες με τις νήσους Φίτζη και τον Ειρηνικό. Ε, είναι λίγα τα χρήματα που διοχετεύονται σε αυτήν την συμφωνία και τα λιεύματα πολλούνται σε, στην αγορά των Βρυξελών, αν πολλούνταν ε, στην ε, ε, αγορά των Βρυξελών, θα, είχαν μια, θα συνιστούσαν αύξηση 6.000% σε σχέση με αυτά που δίνουμε σε αυτές τις χώρες. Οπότε πραγματικά δηλαδή είναι ληστρική συμφωνία για την Πρινσία. Δίνουμε περίπου 480.200 ε, ισοδύναμα. Αν, δώσουμε, αν δούμε σε επίπεδο τόνου είναι 69 ευρώ ένας τόνος τόνου. Δεν χρειάζεται να είμαστε διαστημικοί φυσικοί για να υπολογίσουμε το κόστος του τόνου στα ψαράδικα ε, εδώ στις Βρυξέλλες που είναι 35 ευρώ το κιλό. Ένας τόνος λοιπόν τόνου θα στοιχίζει 35.000 ευρώ ο τόνος. Και εμείς δίνουμε στους ανθρώπους εκείνους 69 ευρώ τον τόνο. Απίστευτα πράγματα. Γιατί δεν ξέρουν τι κάνουμε αυτές οι χώρες για να μας πούνε να πάμε να φύγουμε μακριά. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις, βλέπουμε τις αλληλευτικές συμφωνίες και καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε μόνο. Ε, η γνωμοδότηση αυτή δεν θα περάσει, θα αποφοπλιστεί από την Επιτροπή Αλίας. Αλλά πραγματικά όλα αυτά ε, είναι άδικα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τίποτα άλλο από αλληλεία και λίγο τουρισμό. Τίποτα άλλο δεν έχουν. Ε, πρέπει να είμαστε πιο δίκαιοι απέναντί τους. Δεν μπορεί δηλαδή να τους με 559 ε, ευρώ παίρνοντας ε, οι 559.000 παίρνοντα ε, ε, αλλιεύματα αξίας πολλών εκατομμυρίων από τα ύδατά του. Ε, θα πρέπει επίση να τους δώσουμε τη δυνατότητα να φτιάξουν κάτι, ε, ε, ίσως κονσερβοποιία. Κοιτάζοντας αυτές τις αλλιευτικές συμφωνίες βλέπουμε ότι γίνονται όλο και πιο εξωφρενικές. Εδώ έχουμε μια μεγάλη παρατυπία και γι' αυτό τα, το έθεσα κάπως ομά το θέμα στην έκθεσή μου. Κυρία Μπέρμαν, έχετε ζητήσει το λόγο και μετά ο κύριος Γκέρενς. Ένα διαδικαστικό, κυρία Πρόεδρε. Ορίσαμε συνάντηση των συντονιστών. Έχουμε σημεία άκρο σημαντικά και πολιτική σημασία στην ημερήσια διάταξη που δεν συζητούνται εδώ και μήνες. Σας εκφράζω λοιπόν ε, τις ανησυχίες μου για το πώς ένα τόσο σημαντικό σημείο όπως αυτό που τώρα συζητούμε, υπό πίεση χρόνου συζητιέται. Κοιτάξτε, Μπορούμε να το κάνουμε στις 7 Φεβρουαρίου. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι μας μένουν 15 λεπτά. Μετά δεν θα έχουμε πλέον διερμηνία. Είναι άκρο σημαντικό Και βλέπουμε από άλλα θεσμικά όργανα να δεχόμαστε πιέσει ιδίω από τη ρέλεξ να αποφύγουμε να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα, ενώ σε τρικυμισμένα νερά ψαρεύουμε. Λοιπόν, ως συντονιστές θα πρέπει κάποια απόφαση να λάβουμε. Ζητώ τη συζήτηση αυτή από τον Νοέμβριο. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να συζητούμε περί ανέμων και υδάτων χωρί να μπαίνουμε στην ουσία. Πρόεδρο, δεν είμαι ταχυδακτηλουργό και εγώ, έχω ένα τέταρτο στη διάθεσή μου. Σα λέω λοιπόν, αν θέλετε να δούμε το σημείο 1 ή να δούμε το σημείο αυτό ω πρώτο σημείο στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν μπορώ υλικά και χειροπιαστά να παρατείνω τη συζήτηση. Μα δεν το λέω για εσά, το λέω για όλου μα. Είμαστε συλλογικώ υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή αυτή τη συνεδρίαση. Θα πρέπει όλοι να λάβουν γνώση, να το πούμε στην Προεδρό μας και στην επόμενη συνεδρίαση να είμαστε αυστηρότεροι με το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα δεν θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο. Ε, δεν γίνεται. Εγώ ευχαρίστω να μείνω στις Τρει, Αλλά δεν θα έχουμε πλέον ε, την υποδομή. Κύριε Μπέρμαν για το σημείο περιαλίας. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο ότι έπρεπε να το είχαμε συζητήσει αυτό και στους συντονιστές. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Θα έπρεπε την ερχόμενη εβδομάδα έστω το συντομότερα. Στην ερχόμενη συνάντηση των συντονιστών έστω. Και να αφήσουμε όλα τα άλλα κατά μέρο. Τώρα, κύριε Ντέβα, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Το πρόβλημα της αλίας, όπως πολύ σωστά το θέσατε, είναι θέμα κλοπής. Έχουμε τη συνθήκη με το μέρος μας, τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία απαιτεί να είμαστε συνεπείς και να υπάρχει συνεκτικότητα στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η αλληλευτική μας πολιτική δεν μπορεί να αντιφάσκει με τους στόχους που έχουμε θέσει στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Είναι δική μας υποχρέωση. Είναι υποχρέωση βάση τη συνθήκη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διοργανώσουμε μια κοινή εκδήλωση με την Επιτροπή Αλία και να συζητήσουμε το τι εννοούμε με την συνεκτικότητα. Για αυτό το πολύ συγκεκριμένο σημείο και γενικότερα όμω. Τι πιστεύετε. I would love to do this, but as long... Να το κάνουμε αυτό. Αλλά να μην περιοριστούμε μόνο σε λόγια. Θα πρέπει να πιστούν Χρειάζεται και η γνώμη των νομικών υπηρεσιών για το πώς θα μπορέσουμε να τα περάσουμε αυτά σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφέροντα. Αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά αν είμαστε σοβαροί. Είναι ελάχιστα τα χρήματα που δίνουμε και που όμως επηρεάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον ειρηνικό. Πρέπει λοιπόν να μας πει και η γραμματεία, η γραμματεία μας πώς βάσει συνθήκες της Λισαβόνας, όπως είπε ο κυρίος ε, Μπέρμαν, θα νομοθετήσουμε περισσότερα βάσει της συνοχής. Αν η συνοχή απαιτεί πολιτική συγκεκριμένη για την ανάπτυξη που περιλαμβάνει την αλληλεία, τότε θα πρέπει να περιορίσουμε αυτά που κάνουμε για την αλληλεία τρίτων χωρών, βάζοντας την προτεραιότητα μάλλον στην ανάπτυξη παρά στις αλλιευτικές μας ανάγκες. Χρειάζεται όμως ε, η γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία, το λέω στη γραμματεία, στη Λίντια, ούτως ώστε να βρει μια βάση νομική για να γίνει η συζήτηση με την Επιτροπή Αλίας. Αλλιώς θα μας ακούσουν απλώς και μετά θα συνεχίσουν ε, αταλάντευτοι σε αυτό που κάνουν. Εάν μπορώ να πω την προσωπική μου άποψη, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτή τη συζήτηση, διότι πραγματικά εδώ πηγαίνουμε κάπως ε, ανάποδα ε, στην ανάποδη κατεύθυνση. Δηλαδή και την Επιτροπή μας φορά και την Επιτροπή Αλίας. Θα είναι απόφαση των συντονιστών. Θα πρέπει να το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντησή τους, γιατί το βρίσκω ιδιαίτερα σημαντικό. Συμβαδίζουν οι αποφάσεις των δύο αυτών επιτροπών. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο πολύ σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μάρεκ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στην παρουσίαση της συμφωνίας γιατί ήδη πολλές πληροφορίες ακούσατε και υπάρχουν και στην έκθεση σχετικά με τη συμφωνία. Στηριχθήκαμε στην εντολή του Συμβουλίου, το νέο πρωτόκολλο μονογραφήθηκε στις 7 Μαΐου του 2010 και εδώ τα βασικά σημαντικά στοιχεία του νέου πρωτοκόλλου είναι ότι έχουμε σαφή διάκριση μεταξύ της αναπτυξιακής διάστασης και της ε, συμβολής στην πρόσβαση. Δεν θα επαναλάβω τα νούμερα που ακούσαμε, ίσως διευκρινιστικά υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές με την έκθεση για τη θέση του πρωτοκόλλου. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία επικύρωσης και δεν έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο και από τις δύο πλευρές, οπότε τυπικά δεν ισχύει, αλλά θα γίνει αυτό τους επόμενους μήνες σύντομα. Για την δημοσιονομική συμβολή μας, α, εδώ έχουμε διαφορά από το παρελθόν και έχουμε αυτή τη σαφή διάκριση, ώστε οι 4.480 οι 408 μάλλον 1.200 ευρώ ε, και οι 69 είναι, ανατόνο είναι για την πρόσβαση και τα υπόλοιπα είναι 150.800 ευρώ για τη στήριξη της αλληλευτικής πολιτικής. Επίσης, χθες κατά την παρουσίαση της συμφωνίας με τις ε, νήσους Κομόρες ε, τονίστηκε ότι δεν είναι, μόνο, δεν είναι αναπτυξιακές συμφωνίες, είναι το κομμάτι της αλίας και το κομμάτι της ε, ανάπτυξης και τα δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέσον όρο για τα λιεύματα τόνου το 69 ε, έχουμε 65-35 αναλογία μέχρι τώρα, αυτή είναι μια μικρή διόρθωση και επίσης δεν πληρώνουμε για τον τόνο αλλά η τιμή αυτή και πώς διαρθρώνεται στη συμφωνία στηρίζεται στην πρόσβαση. Δηλαδή έτσι μπορεί να υπάρξουν ελιευτικές δραστηριότητες από τους στόλους μας και μετά η δομή των τιμών στις αγορές καθορίζεται από τις διάφορες αγορές, στα διάφορα επίπεδα. Αυτό αφορά τη διάρθρωση των τιμών. Επίσης, πολύ σύντομα να πω και για κάποια άλλα θέματα που αναφέρεται στην έκθεση. Το ένα αφορά τα αλλιεύματα και τις διαδικασίες. Θα ήθελα να πω ότι οι διαδικασίες και η επαλήθευση των αλλιευμάτων γίνεται από Επιστημονικό Ινστιτούτο και επίσης ε, μια άλλη νομική υποχρέωση στηρίζεται στον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο που επιβάλλει στα κράτη-μέλη ε, την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ότι ε, είναι οι πυλώνες ε, για τα αλλιεύματα. Τώρα για τους μηχανισμούς καθ' αυτούς ε, έχουμε ακαιρεότητα, διαφάνεια όπως και κατά το παρελθόν. Τώρα προσθέσαμε και κάποιες νέες ρήτρες αναθεώρησης. Το ένα είναι της αναστολής της δημοσιονομικής συνεισφοράς στην τομεακή πολιτική αν δεν υπάρχει συμμόρφωση προς την πολιτική. Οπότε θα πρέπει να ε, έχουμε έτσι μια διασφάλιση, μια εγγύηση ότι θα παρακολουθούμε λεπτομερέστερα τα θέματα. Επίσης συμφωνήσαμε με ότι θα πρέπει οι τοπικές συνθήκες να γίνονται σεβαστές και στη Μικρονησία. Δηλαδή υπάρχουν και σε περιφερειακό επίπεδο κάποιες προϋποθέσεις ε, και δεσμεύσεις. Τώρα, οι συνθήκες για τους ε, ε, τοπικούς αλληλείς θα προσπαθήσουμε βέβαια να ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας κατά τις κοινέ συναντήσεις, συνεδριάσεις, να θέσουν τα θέματα αυτά ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να εξεταστούν. Αυτές είναι οι πληροφορίες με βάση τις εκθέσεις και ε, ε, χαιρόμαστε για την έκθεση. Προσπάθησα να είμαι σύντομος, αλλά αν υπάρχει ε, ενδιαφέρον από κάποιο κράτος μέλος ή κάποιο αξιότιμο βουλευτή, μπορούμε να συζητήσουμε για την Ελευθερική Συμφωνία περισσότερο. Ο κύριος Ντέβα τώρα για, να, για τα συμπεράσματα. Συγγνώμη, δεν θέλω να είμαι προσβλητικός, δεν θέλω να είμαι αγενής, συνήθως είμαι ευγενής. Προσπάθησα να παρακολουθήσω αυτά που λέτε, αλλά δεν βγάζουν νόημα. Ούτε απαντάτε στις ερωτήσεις ε, της ε, έκθεσης. Μας είπατε κάποια τεχνική ορολογία, ελπίζοντας ότι θα καταλάβουμε εγώ. Σας καλώ να έρθετε μαζί μου σε μια συνέντευξη τύπου και να εξηγήσετε στο, στα ΜΜΕ ακριβώς τι είναι αυτά που κάνουμε εκεί στη Μικρονησία και πώς ε, ε, νομιμοποιούμεθα να πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε στον κόσμο εκεί. Αν είστε πρόθυμος για κάτι τέτοιο, εγώ θα γράψω επιστολή στον κύριο Μπαρόζο και θα του τα εξηγήσω όλα αυτά και θα του πω ότι θέλω να αξιωματούχο της Κομισιόν σε κοινή μαζί μου press conference για να εξηγήσουμε στην, στον τύπο, στα ΜΜΕ, τι ακριβώς κάνουμε στην Μικρονησία. Ευχαριστούμε κύριε Ντέβα. Νομίζω ότι έχουμε πει όσο έπρεπε να πούμε. 3 Μαρτίου θα ψηφιστεί. Ε, στις 7 Φεβρουαρίου, στις 6 λίγη προθεσμία για την υποβολή των πολιών. Άλλε παρατηρήσει ο κύριο Γκέρεν. Ναι, επειδή δεν μπορέσαμε να κάνουμε τη συνάντηση των συντονιστών σήμερα, θα ήθελα παρόλα αυτά να επανέλθω στην πρόταση που γίνεται στο έγγραφο από τη Γραμματεία. Νομίζω ότι θα είναι απαραίτητο να ορίσουμε πολύ γρήγορα, να έχουμε μάλλον πολύ σύντομα συνάντηση με τον διευθυντή της ΔΕΦΚΟ. Αμέσως, αμέσως να έρθει να μας δει, να το αποστείλει με πρόσκληση. Συμφωνούμε. Στηρίζω την ε, αίτηση του κυρίου Γκέρενς, λέει ο κύριος Μπέρμαν. Πολύ ωραία, το σημειώνουμε. Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες 7 Φεβρουαρίου. 3 με 6.30. Ελπίζω ότι θα είμαστε όλοι εδώ. Η συνεδρίασή μας ε, λίγη. Σας ευχαριστώ όλους και όλες.